όπως είπαμε και πριν βεβαίως η συμβάση της ΔΟ είναι μέρος της βασικής κοινωνικής πολιτικής μας. Κυρώνοντας τη συζήτηση αυτή θέλω να σας αναγγείλω ότι έχω λάβει τρεις προτάσεις ψηφίσματος. Η μία πρόταση είναι από κοινού από την ε, ε, ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και την ομάδα των Φιλελευθέρων με την ομάδα της Αριστεράς. Η άλλη πρόταση είναι από την ε, ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και η τρίτη από τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές η συζήτηση έληξε εδώ και η ψηφοφορία θα γίνει αύριο για το θέμα αυτό. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια μας διάταξη είναι η δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την παγκόσμια διάσκεψη του Διεθνούς Οργανισμού Τροφίμων και Διατροφής με θέμα την επισητιστική ασφάλεια και την εξάλληψη της πείνας από τη γη. Θα ξεκινήσουμε με την δήλωση της Επιτροπής. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Uh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριοι βουλευτές, το, η Παγκόσμια Σύνοδος Κορυφής της περασμένης εβδομάδας στο Ιρόμι είναι μία από τις πολλές εκδηλώσεις που οργανώνονται φέτο τον Ιανουάριο στην Μαδρίτη, μετά στη Λακουίλα, μετά στην Νέα Υόρκη κτλ. Η βασική αρχή όλων αυτών των εκδηλώσεων ήταν ότι συνειδητοποιούμε πως δεν πως αποτυγχάνουμε να αντιμετωπίσουμε την πείνα παγκοσμίω και χρειάζεται να περισσότερη προσπάθεια σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες τα πράγματα επιδεινώνονται και λόγω της κλιματικής αλλαγής που δημιουργεί επιπλέον προκλήσεις για τις χώρες αυτές που δεν μπορούν να είναι αυτάρκες ή να έχουν την ε, απαιτούμενη επιστηστική ασφάλεια. Τους τελευταίους μήνες τα πράγματα επιδεινώνονται πραγματικά και η ασφάλεια επιστηστική έγινε και πάλι επίκαιρη. Όμως Τώρα πρέπει να τελειώνουν τα ωραία λόγια, τώρα πρέπει να αποδειθούμε σε δράσεις και πρέπει να καταφέρουμε αυτό που ορίστηκε σαν πρώτο στόχο της χιλιετίας να ε, ε, έχει καταπολεμηθεί κατά το ίμιση η πείνα μέχρι το 2015 αυτό το χρειάζεται, αυτό πρέπει να γίνει πραγματικότητα. Επίσης υποσχεθήκαμε ότι πρέπει να υπάρχει ένας καλός συντονισμός μέσω μιας επιτροπής για την επιστημιστική ασφάλεια ε, και η επιτροπή αυτή είναι μια ε, βασική συνιστόσα για την όλη δουλειά που θα γίνει στον τομέα της γεωργίας και της, ε, της διατροφής. Εδώ η σύσταση αυτής της Επιτροπής και ο συντονισμός μέσω της Επιτροπής αυτής είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα το οποίο θα γίνει και που θα βασίζεται στα, σε επιστημονικά στοιχεία και όπου θα συμμετάσχουν και ο ιδιωτικό και ο δημόσιο τομέα και μη κυβερνητικοί οργανισμοί. Το σύστημα ελπίζουμε ότι θα γίνει πιο αποτελεσματικό από ότι είναι. Τρίτη υπόσχεση που δόθηκε είναι να βελτιωθεί η χρηματοδότηση για όλου αυτού του πολύ σημαντικού τομεί. Αν θέλουμε να επιτύχουμε τον πρώτο στόχο τη χιλιετία, να ε, καταπολεμηθεί κατά το ίμιση πείνα μέχρι το 2015, τότε πραγματικά πρέπει να γίνουν σεβαστές κάποιες υποσχέσεις που δόθηκαν από όλους για την ε, επιδότηση αν θέλετε του όλου αυτού προγράμματος 0,7% του ΑΕΠ ε, η, πέρα από την ε, πέρα από το τι γίνεται και τι πρέπει να κάνουμε σχετικά με την ανάπτυξη σε χώρε. χώρες δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ε, ότι έχουν ήδη ληφθεί κάποιες αποφάσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν σεβαστέ και ε, να εφαρμοστούν η, Υπάρχει ήδη η Food Facility. 85% των κονδυλίων αυτών έχουν ήδη δεσμευτεί μέχρι το 2011 από εκεί και πέρα για να μπορέσουμε να ε, εφαρμόσουμε τις υποσχέσεις μας θα πρέπει να αναπτύξουμε επίσης ειδικού δείκτες, ειδικά benchmark και ειδικού μηχανισμούς ελέγχου για να ελέγχουμε τις επενδύσεις που γίνονται προς την κατεύθυνση των στόχων μας και θα πιστεύουμε ότι ακόμη και αν οι δωρητές δώσουν μεγάλα ποσά δεν θα μπορέσουν να επιτύχουν τίποτε αν τα κράτη-μέλη δεν κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν στον τομέα της γεωργίας. Η επιστημιστική ασφάλεια επίσης όταν συζητείται ε, χρησιμοποιεί κάποιους όρους οι οποίοι πρέπει να χρησιμοποιούνται με φιδό και σωστά. Η αυτάρκεια, η αυτονομία είναι όροι που δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εύκολα. Θέλουμε όλοι να έχουν πρόσβαση στην τα τρόφιμα. Ε, εδώ μπαίνουμε στα χωράφια της ένδυας και της καταπολέμησης της ένδυας. Από εκεί και πέρα θέλουμε να υπάρχει πρόσβαση σε φτηνότερα τρόφιμα. Εκεί μπορούμε να επέμβουμε στις τιμές. Η οποιαδήποτε στρατηγική βεβαίως, σαν και αυτή προσπαθούμε να εφαρμόσουμε τώρα, δεν θα χρειαζόταν νέα ναι, αγορές, λειτουργούσαν καλά, αλλά δεν λειτουργούν. επίσης, ο γύρος της Ντόχα ε, αν είχε καταλήξει σε σωστά αποτελέσματα ίσως θα είχε βοηθήσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιτελέσει κάποια πρόοδο αν θέλετε η οποία όμως δεν αρκεί. Η διαδικασία PCD πρέπει να συνεχιστεί. Η κοινή η αγροτική πολιτική στην εξωτερική πτυχή της έχει επηρεάσει επίσης τα πράγματα και στο εσωτερικό έχει βοηθήσει τους αγρότες να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την παγκοσμιοποίηση αν θέλετε που δημιουργείται μέσω των γύρων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου πιστεύουμε ότι υπάρχουν όμως και άλλα προβλήματα όπως παραδείγματο χάρη σε αναπτυσσόμενες χώρες όπως χώρες ΑΚΕ για τις οποίες είναι εν μέρη υπεύθυνη ή μπορεί να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουμε ότι πρέπει να βοηθήσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες για το θέμα αυτό και όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και οι άλλες χώρες και οι άλλες περιοχές του πλανήτη. Αν θέλ, επανέρχομαι στο στόχο μας για την καταπολέμηση της πείνας κατά το ίμιση μέχρι το 2015. Για να γίνει αυτό πρέπει να ενισχυθούν οι επενδύσεις στον τομέα της γεωργίας και να τηρηθούν κάποιες βασικές αρχές. Πάρουν ομιλητές εξ των πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Ντές για δύο λεπτά εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Mr. Ντές, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, για μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πολύ σημαντικό να ασχολούμεθα με το θέμα της πείνας στο πλανήτη μας. Δεν μπορούμε να αγνοούμε το γεγονός ότι πολλοί πεινούν και μεταξύ αυτών είναι πολλά παιδιά που πεινούν. Θυμούμε ότι παλιό και παλιότερα διεθνείς οργανισμοί, ΟΗΕ, Διεθνή Παγκόσμια Τράπεζα και τα λοιπά έκαναν διάφορες ε, δηλώσει στο παρελθόν που έλεγαν ότι η πείνα θα καταπολεμηθεί, δεν θα υπάρχει πείνα στο μέλλον. Αντιθέτως η πείνα αυξήθηκε και η κατάσταση επιδεινώθηκε. Γιατί υπάρχουν πολλοί λόγοι, υπάρχουν χώρες όπου φταίνει οι κυβερνήσεις στο Ζιμπάμπουε παραδείγματος χάρη η κυβέρνηση και ε, ε, οι κομμουνιστές κατάφεραν να δημιουργήσουν μια κατάσταση κατά την οποία ο πληθυσμός πεινά αλλά φταίμε και εμείς, φταίμε και εμείς γιατί δεν μα, διότι προσπαθούμε να κάνουμε, να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές με προοπτική πεντηκονταετίας ή εκατονταετίας ο άνθρωπος που πεινάει δεν ενδιαφέρεται για σχέδια που με προβολή στο μέλλον ενδιαφέρεται να φάει σήμερα και το αυτό το να αναφέρεται ότι μέχρι το 2050 θα πρέπει να καταπολεμηθεί με κατά το ίμιση η πείνα είναι υπερβολικό για μένα νομίζω ότι ε, ο, οι άνθρωποι αυτοί που πεινούν σήμερα δεν θα ζουν μέχρι ε, τότε Ευχαριστώ κύριε Ντές για την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ο κύριος Κάπουλα Σάντος για δύο λεπτά Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Τα αριθμητικά στοιχεία που καταδεικνύουν την ε, ένδια, την πείνα στον κόσμο είναι τόσο δραματικά που είναι σχεδόν επέσχυντο να τα αναφέρουμε. Το πιο ιερό από τα δικαιώματα καταστρατηγείται, το δικαίωμα στη ζωή, στην αξιοπρέπεια και όχι σε μια καθημερινή πάλι για επιβίωση. Η καταπολέμηση της πείνας θα πρέπει να είναι η προτεραιότητα των προτεραιοτήτων όλων των πολιτικών ε, προγραμμάτων. Και γι' αυτό θα πρέπει να κινητοποιηθούν όλοι οι δυνατοί πόροι. Δυστυχώς γνωρίζουμε ότι οι πόροι συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών δεν είναι ε, πάντα το μεγαλύτερο εμπόδιο. Το πρόβλημα είναι η διαχείριση και η χρήση των πόρων και η απουσία μιας αποτελεσματικής ε, συλλογικής προσπάθειας ενός συντονισμού σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό επίπεδο. προτείνουμε στο ψήφισμά μας κάποιες συστάσεις που αν ακολουθηθούν μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά πιστεύω στην άμβλυνση αυτού του προβλήματος. Γι' αυτό απευθύνω έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει το ψήφισμα και να προτείνει μέτρα και διαδικασίες που θα τις μεταφράσουν αυτές τις εξαγγελίες στην πράξη. Οι οικονομικές και πολιτικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε είναι και μια ευκαιρία αλλαγής της πολιτικής ε, της Ευρωπαϊκής Ένωση στον τομέα. Η κοινή αγροτική πολιτική, η κοινή ελληνική πολιτική, των οποίων η εκβάθρον μεταρρύθμιση θα ξεκινήσει με τα νέα με τις νέες αρμοδιότητες που έχουμε από τη συνθήκη της Λισαβόνας είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να περάσει από τα λόγια στις πράξεις. Οι Ευρωπαίοι σοσιαλιστές είναι, κινητοποιούνται προς αυτή την κατεύθυνση και ευχόμεθα η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι λοιπές πολιτικές ομάδες να μας συνοδεύσουν σε αυτή την αποστολή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και συνάδελφε. Ο κύριος Λίον για 1,5 λεπτό παρακαλώ από την ομάδα των φιλολευθέρων. Uh, thank you, uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους ε, που ήδη συνέβαλαν. Το πρώτο που θα ήθελα να πω είναι το, οι τιμές των, ε, των ε, τροφίμων μας δείχνουν ακριβώς το γεγονός ότι διπλασιάστηκαν δηλαδή οι τιμές του ρυζιού για παράδειγμα και υπήρχε μια δυσανάλογη συνέπεια σε φτωχούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Μας δείχνει ήδη πολλά πράγματα. 75 εκατομμύρια άτομα περισσότερα θα αρχίσουν να πεινούν επειδή αυξήθηκαν πάρα πολύ τιμέ το 2007 και το 2008. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Και πολλές χώρες ε, είδαμε ότι υπήρξε και πολιτική αστάθεια λόγω της ε, ραγδαίας αύξησης των τιμών. Επειδή θα φτάσει τα 9 δισεκατομμύρια ε, ο πληθυσμό του πλανήτη, θα έλεγα ότι η επιστημιστική ασφάλεια είναι ένα σημαντικότατο ζήτημα το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπίσουμε το συντομότερο δυνατόν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει τι αναπτυσσόμενε χώρε ε, για ε, βιώσιμες, ε, βιώσιμη γεωργία και να μπορούν να έχουν αυτάρκεια στα τρόφιμα ε, όπως είπε και η Επιτροπή στη δήλωσή της, ε, και να υπάρχει και μία αναγνώριση ότι η Ευρώπη έχει κάνει πάρα πολλά ως προς την ε, απελευθέρωση των αγορών. Ένα από τα πολλά προβλήματα των αναπτυσσομένων χωρών είναι η ανεπάρκεια του πολιτικού συστήματος, η ανεπάρκεια των κυβερνήσεων να μπορέσουν να δημιουργήσουν ένα σταθερό νομικό σύστημα που δίνει τη δυνατότητα στους αγρότες να αξιοποιήσουν τα ωφέλη των τιμών της αγοράς. Επειδή θα, αυξηθεί ακόμη περισσότερο, θα αυξηθούν ακόμη περισσότερες, περισσότερο οι τιμές και επειδή η Γεωργία έχει πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει, πιστεύω ότι πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να συμμετέχουμε στην επιστημιστική ασφάλεια στο μέλλον. Έχει το λόγο για δύο λεπτά. Madame la Présidente, euh, Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, ο ΦΑΟ δεν ε, κατάφερε να αντιμετωπίσει μια μεγάλη πρόκληση το περασμένο Σαββατοκύριακο και κρίμα. Ε, πάρα πολλοί άνθρωποι υποφέρουν από πείνα, 40 εκατομμύρια παιδιά ε, και γυναίκες πεθαίνουν από την πείνα κάθε χρόνο. Έχει αυξηθεί ο το, ο αριθμός αυτός από το 1996 και η κοινωνική κρίση ε, ε, ε, επιδίνωσε ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Οι χώρες του Νότου είναι τα πρώτα θύματα της όλης κατάστασης. 10% της, ε, του προπολογισμού της διαφήμισης θα έδινε την απαραίτητη υποστήριξη στις αναπτυσσόμενες χώρες για να μπορέσουν να ε, επενδύσουν σε υποδομές γεωργικής φύσεως. Γιατί η επιστηστική ασφάλεια είναι μια βασική απειλή που, δημιουργεί, που αποτελεί μια, είναι απειλή και για την ειρήνη. Ε, το 2050 θέλουμε να μειώσουμε ε, την ε, ένδια. Υπάρχει όμως το θέμα της διάβρωσης του εδάφους, υπάρχει το θέμα των εκπομπών αερίου θερμοκηπίου, υπάρχουν τόσα πολλά προβλήματα και που μας θέτουν σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση και πολύ ευαίσθητη, πολύ πιο ευαίσθητη από ό,τι πριν από 40 χρόνια. Η εξάρτηση, η φτώχεια, ε, η εξάρτηση από τις εισαγωγές είναι ένας από τους βασικούς λόγους ε, της έλλειψης επιτιστικής ασφάλειας. Είναι σημαντικό να υπάρχει παραγωγή σε τοπικό επίπεδο. Από τα τέλη της δεκαετίας του 50 η Ευρώπη έχει μια κοινή γεωργική πολιτική για να παράγει τα τρόφιμα τα οποία χρειάζεται για να μπορέσει να προστατεύσει ε, την εσωτερική της παραγωγή και να προστατεύσει τους καταναλωτές της. Αυτό το, αυτό, αυτή η αυτονομία, αυτή η επισητιστική κυριαρχία ε, είναι, πρέπει, να, πρέπει να είναι κάτι ε, που, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση όλες οι χώρες του κόσμου. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Thank you very much, uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ψήφισμα έχει να κάνει με τη δυτή πρόκληση και της πείνας και της φτώχειας ε, για μεγάλο τμήμα του πληθυσμού και για την επιστημιστική ασφάλεια στο μέλλον. Έχουμε μπροστά μας την εξή κατάσταση. Από τη μία αυξάνεται ο πληθυσμός, από την άλλη είναι πρόκληση η παραγωγή τροφίμων λόγω της κλιματικής μεταβολής και λόγω της αύξησης του κόστου της παραγωγής των τροφίμων. Ε, το θέμα της γεωργικής πτυχής ε, που έχει να κάνει με την επιστημική ασφάλεια είναι σημαντικός παράγοντας επίλυσης του προβλήματος, αλλά θα έπρεπε να επικεντρωθούμε και στην καλή ε, διακυβέρνηση στις διάφορες χώρες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν θέλουμε να είμαστε επιτυχείς στην αντιμετώπιση της πείνας, όπως για παράδειγμα ανέφερε προηγουμένως ο κύριος Ντες, στην Σιμπάμπουε για παράδειγμα, κάποτε μπορούσε να ε, τρέφεται χωρίς πρόβλημα, αλλά μετά από την κατάσταση που δημιούργησε ο Μουγκάμπε τα πράγματα είναι δραματικά και δεν γίνεται πια αυτό. Ε, οι αναστατώσει που υπάρχουν, η όλη αστάθεια που θα προκύπτει από αυτό δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχε το πρόβλημα της επιστημικής ασφάλειας. Ευχαριστώ. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση ήθελε να παίξει έναν ε, θετικό ρόλο ε, στον κόσμο, αν θα έπρεπε να δείξει έναν νέο ανθρωπισμό, θα έπρεπε να ακούσει την κοφαντική φωνή, ε, την εκοφαντική φωνή όλων αυτών των ανθρώπων που υπουνούν. Εμεί εδώ κάνουμε πολύ ωραίου λόγου, λέμε πολύ ωραία πράγματα, αλλά θα έπρεπε να. Πώ μπορούμε να έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μα όταν κάθε πέντε δευτερόλεπτα πεθαίνει ένα παιδί από την πείνα στον κόσμο έχουμε αυτό τον άκρατο φιλελευθερισμό που δημιουργεί αυτό το μεγάλο πρόβλημα στο σημερινό κόσμο. Δεν μπορούμε πια να θρέψουμε τον κόσμο και το καπιταλιστικό σύστημα ε, δημιουργεί καθιστά ουσιαστικά τα τρόφιμα εμπόρευμα και γι' αυτό ακριβώς πρέπει να αλλάξουμε ε, ριζικά την πολιτική μας και να υποστηρίξουμε τη ΦΑΟ, το ΦΑΟ και να, τους δώσουμε, του δώσουμε τα μέσα να επιτύχει όλα αυτά που θέλουμε. Για να περάσουμε στην πράξη, το, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να ζητήσει το σεβασμό ε, των σχετικών αρχών από όλα τα κράτη, ε, αποζημίωση επίσης με εγγυημένο μισθό όλων των γεωργών, να γίνουν σεβαστοί επίσης, ε, να γίνουν σεβαστές ε, οι ίδιες δεσμεύσεις και για τις αναπτυσσόμενες χώρες, ε, να μην αγοράζουν πια τις γέες οι πολυεθνικές και να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι τα τρόφιμα δεν μπορεί να είναι ένα εμπόρευμα του ΠΟΕ μόνο. Πρέπει να ακούσουμε αυτή την εκοφαντική κραυγή της πείνας και αυτό θα έκανε την Ευρώπη πολύ πιο σημαντική. Τώρα για δυόμιση λεπτά ο κύριος Μπέλντερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα δέκα χρόνια που είμαι βουλευτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχω ε, ακούσει πολλά μεγάλα λόγια. Και ο πρόεδρος Μπαρόζο χρησιμοποίησε μεγάλα λόγια, μας είπε ότι αποτύχαμε στον αγώνα κατά της πείνας. Αυτό είναι σκάνδαλο. Είναι ένα στίγμα που όλοι φέρουμε τέλος της παράθεσης. Κοιτάξτε, το αποτέλεσμα όντω είναι απογοητευτικό. όχι μόνο οι άνθρωποι πεινούν παγκοσμίω, αλλά και όσοι μπορούν να κάνουν κάτι δεν το κάνουν η χρήση ας πούμε γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή βιοεθανόλης ε, επιτείνει το πρόβλημα της πείνας. Δεν θα πρέπει να πρημοδοτούμε αυτές τις πρακτικές. Πώς θέλετε χώρες ε, στην ε, Αφρική ή στον Τρίτο Κόσμο γενικότερα να παίρνουν βοήθειες αλλά συγχρόνω να μην μπορούν να παράγουν τα δικά του τρόφιμα γιατί τα όσα λίγα παράγουν τα κάνουν καύσιμα για να κινούνται τα αυτοκίνητα. Είναι και οι αναπτυσσόμενε χώρες θέλω να πω κάπως υπεύθυνε. Εγώ ξεφίλησα την ε, τελική ε, δήλωση αλλά και άλλα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γίνεται πάντα λόγος ε, ε, για την προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε, για την ηθική μας υποχρέωση, αλλά θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι ε, δεν έχουμε κάνει και πολλά. Μόνο λόγια και εξαγγελίες και ο κόσμος, ο κοσμάκης, τολμώ να πω, θέλει να γεμίσει την κοιλιά του. Αυτό είναι το πρόβλημά του. Εγώ ε, προσωπικά ε, θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ για να το επιτύχω. Εγώ από τους μη για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμμετέσχα πρόσφατα ε, στην διάσκεψη κορυφής της ΦΑΟ και έμαθα από πρώτο χέρι πώς έχουν τα πράγματα θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι οι υποσχέσεις και τα παχιά λόγια που είναι το αποτέλεσμα αυτών των ε, ε, διασκέψεων κοστίζουν χρήματα για να οργανωθούν αυτές οι συνδιασκέψεις ε, και αυτές οι υψηλού επίπεδου συναντήσεις δαπανώνται εκατομμύρια εκατομμυρίων. Αν είχαν χρησιμοποιηθεί αυτά τα εκατομμύρια για να δοθεί επιστηστική βοήθεια στους ανθρώπους που πεθαίνουν από την πείνα δεν θα είχαμε τόσο μεγάλο πρόβλημα. Η χώρα μου έχει το πιο γόνιμο έδαφος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Βούλγαροι Γεωργοί θα μπορούσαν να δώσουν, ε, έδιναν φαΐ στις πιο πυκνοκατοικημένες ε, περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Όλα αυτά όμως τελείωσαν. Οι ποσοστώσεις που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιβάλει στην Βουλγαρία καταστρέφουν τη γη. Χωματερές έχουμε μία μόνο περιφέρεια της ε, χώρας μπορεί να παράγει το σύνολο της ποσόστοσης που έχουμε για το συγκεκριμένο προϊόν. Πώς θέλετε να τα βγάλουμε πέρα έτσι. Πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για εξορθολογιστική ε, παραγωγή και για ε, κάλυψη των αναγκών μιας χώρας ευρωπαϊκής και μάλιστα της ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι δυνατόν να γίνουν αυτά από τους γραφειοκράτες των Βρυξελών. Τον κατάλογο των ομιλητών, ο κύριος Κατσμαρέκ θα πάρει το λόγο για δύο λεπτά. Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu, Szanowni Państwo. Liczba osób cierpiących głód i Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, πάνω από ένα δις ανθρώπων ζει σε κατάσταση άκρας ένδειας και πείνας. Αυτό δεν είναι όμως το αποτέλεσμα του καπιταλιστικού συστήματος. Υπάρχουν πολύ χειρότερα συστήματα από το καπιταλιστικό. Στην Ευρώπη, για παράδειγμα, πριν από πολλά χρόνια, μια χώρα με πολύ καλές γεωργικές και αγροτικές ε, συνθήκες, ε, η Ουκρανία... Ε, αντιμετώπισε προβλήματα πείνας σε τεράστιο βαθμό. Πολλοί άνθρωποι πέθαναν. Ε, τώρα στον ΟΗΕ ε, πολλά μέλη, ε, πολλές χώρες μέλη του ΟΗΕ ενέκριναν ένα ψήφισμα με συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τους στόχους της χιλιετίας. Πρέπει να διαρωτηθούμε αν είναι ρεαλιστική αυτή η στόχη. Είναι σωστές οι πολιτικές μας, είναι σωστές οι προτεραιότητες μας. Πιο συγκεκριμένα, ε, πόσο πιο σημαντικό είναι η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής από την καταπολέμηση της πείνας. Ερωτώ, αντί να προσπαθούμε να αντιστρέψουμε τις ε, συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, δεν θα ήταν καλύτερο να κάνουμε μια προσπάθεια για να ε, εξαλείψουμε την πείνα στον κόσμο. Αν είχαμε εξαλείψει την πείνα πρώτα, κανείς δεν θα μπορούσε να μας κατηγορήσει ότι έχουμε θέσει λάθος προτεραιότητες και ότι αφήνουμε το γάμο για να πάμε για πουρνάρια όπως ανέφερε ο κύριος Ντες. Η γεωργία είναι πολύ σημαντική και θα είναι ακόμα πιο σημαντική για τα επόμενα χρόνια και θα πρέπει να πείσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες να επενδύσουν οι ίδιες στην γεωργία οι ίδιε οι αναπτυσσόμενε χώρε είπαν ότι θα επενδύσουν 10% του ΑΕΠ του για την γεωργία. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα γίνει αυτό. Είναι ο μόνο τρόπο να ε, αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Ο κύριος Σάριφ, ο επόμενος εγγεγραμμένο ομιλητής, δεν φαίνεται να είναι στην αίθουσα και το λόγο θα πάρει ο κύριο Λουί Μισελ για τρία λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, εκτός από τον κύριο Σίλβιο Μπερλουσκόνη του οποίου η χώρα φιλοξενούσε την διάσκεψη κανένα μέλος ε, της ομάδας των 8 δεν ήταν παρόν ε, στο, στη διάσκεψη κορυφής της ΦΑΟ. Μία άκρος λοιπόν πολιτική συνάντηση με οικονομική, κοινωνική και δημοσιονομική διάσταση κατήντησε μία τεχνική συνεδρίαση. Ο στόχος του κυρίου Ντιούφ ήταν να διασφαλίσει επιστημική ασφάλεια με βιώσιμο τρόπο στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η οικονομική και δημοσιονομική κρίση, το γνωρίζουμε, βεβαίως επιτείνει το πρόβλημα και το οποίο είναι ε, δυστυχώς ε, επίκαιρο παραποτέ. Ένα δις ανθρώπων πεινούν στον κόσμο, το ένα έκτο της, ε, του παγκόσμιου πληθυσμού, 1% παραπάνω από το 2005, 500 εκατομμύρια παραπάνω από το 2008. Κάτι το οποίο, όπως είπε ο κύριος Μποβέ, θα δημιουργήσει νέες μορφές συγκρούσεων ε, ιδιαίτερα ανησυχητικέ. Η έλλειψη επενδύσεων στη Γεωργία οδήγησε σε αυτό το φαινόμενο της επιστημιστική και διατροφικής ανασφάλειας όταν η γεωργία είναι το μόνο μέσο επιβίωσης του 70% του τρίτου, των ανθρώπων του τρίτου κόσμου, ε, πώς είναι δυνατόν να ε, ε, διέλθουμε της κρίσεως και οι εξαγγελίε μας έχουν μείνει κενό γράμμα. Ούτε χρονοδιάγραμμα, ούτε στρατηγική, ούτε πολιτική βούληση υπάρχει από τις ε, πλούσιες χώρες. Πού βρισκόμαστε λοιπόν σε σχέση με τις δεσμεύσεις ε, της ομάδας των 8 ε, Ξέρω τι δυσκολίε που υπάρχουν να κινητοποιηθούν οι δωρητέ, Θυμάμαι ακόμα τη μάχη που δώσαμε και που έδωσε και ο πρόεδρος Μπαρόζο για να ε, πάρει αυτό το ε, ψίχουλο που είναι το 1 δις ευρώ για την λεγόμενη επιστημιστική διευκόλυνση ε, εγώ δεν πιστεύω κύριε Επίτροπε, δεν πιστεύω στη συνταγή του σοσιαλιστή συναδέρφου που βλέπει τον εχθρό στο, στο, τέλος πάντων στο πρόσωπο του καπιταλισμού. Δεν βλέπω ε, πώς ε, θα έχουμε λύση με, αυτές τις, ε, με αυτούς τους αφορισμούς, τους ιδεολογικούς αφορισμούς που δεν προσφέρουν τίποτα. Η πανάπτυξη, ο μαρξιστικός σκοταδισμός έχει πολύ μεγαλύτερη ευθύνη από ότι ο φιλελευθερισμός. Αυτά ήθελα να πω γιατί δεν ήθελα να περάσει αυτή η δήλωση στους κόλπους του Κοινοβουλίου έτσι ελαφρά τη καρδία. Είναι θέμα πνευματικής εντιμότητος. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μισελ. Ο κύριος Αρτζεντίνη για ένα λεπτό έχει το λόγο τώρα.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 Ε, περιέγραψαν το πρόβλημα και την πολιτική πραγματικότητα αλλά υπάρχει μια καινούρια τάση στη γεωργία βιοτρόφιμα, βιομάζα και τα και υπάρχει πέραν αυτού και το περίφημο land grabbing δηλαδή προσπόρηση αν θέλετε γεωργικών γεών αυτό συμβαίνει, συμβαίνει στη Μαδαγασκάρη παραδείγματος χάρη οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι υποχρεωμένοι να καταπολεμήσουν αυτό τον, αυτή τη μέθοδο, αυτό το θέμα, το καινούριο απεικιοκρατικό τρόπο προσπόρηση αν θέλετε. Γιατί δεν έγινε κάτι τέτοιο ήδη. Στην ΚΑΠ εμείς η Ευρώπη ε, παράγει πολύ, πολλά τρόφιμα. Οι Ευρωπαίοι έχουν να φάνε και, και υπάρχουν ε, και μεγάλοι και μικροί αγρότες. Σε άλλες χώρες όμως υπάρχει πρόβλημα και ε, υπάρχει ανάγκη ε, εισαγωγών και σε άλλες χώρες αλλά και στην Ευρώπη. Και η κυρία Άστορφ έχει το λόγο τώρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε και τα Ηνωμένα Έθνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνούν ότι πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη παραγωγικότητα κατά 50% ίσως στον γεωργικό τομέα. Αυτό είναι γεγονός και είναι ένας στόχος ο οποίος πρέπει να επιτευχθεί. Συγχρόνως όμως οι γεωργοί πρέπει να το κάνουν αυτό με λιγότερη γη, με λιγότερα αέρια του θερμοκηπίου, με λιγότερο νερό, με λιγότερη ενέργεια. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε τα εξή. Πρώτα-πρώτα οι κυβερνήσεις πρέπει να επενδύσουν περισσότερο στην έρευνα και την ανάπτυξη. Δεν έχουμε τα στοιχεία επί των οποίων να βασίσουμε ένα σχέδιο για το μέλλον. Δεύτερον, δεδομένης κατάσταση των αγορών, των διεθνών αγορών, χρειάζεται ένα δίκτυο ασφαλείας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τρίτον, η επισητιστική ασφάλεια έχει κόστος, ένα κόστος το οποίο δεν μπορούμε να το μετακυλήσουμε στους καταναλωτές. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ισχύ ισχυρή κοινή αγροτική πολιτική και πρέπει να κερδίσουμε στη συζήτηση για τον προπολογισμό. Τώρα ο κύριος Φερέιρα θα πάρει το λόγο για 1,5 λεπτό. Senhora Presidente, a declaração final adotada na última cimeira da FAO pelos seus 193 e e países membros é infelizmente στην τελευταία σύνοδο κορυφής της ΦΑΟ με πάνω από 150 χώρες ε, ουσιαστικά δεν έγινε τίποτα για την εξάλληψη της πείνας και της φτώχειας. Χρειαζόμαστε κάτι πιο απτό για να μπορέσουμε να ε, καταπολεμήσουμε αυτές τις μάστιγες. Γύρω στα δέκα αν ε, δεν κάνω λάθος, ανά πάσα στιγμή 15 παιδιά ε, πεθαίνουν από πείνα ή από φτώχεια. Ε, αυτά είναι ντροπέ στην ιστορία του πλανήτη που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Όπως είπε και ο κύριος Λούι Μισελ, δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε το παιχνίδι αυτό του άκρα του φιλελευθερισμού. Μπορούμε να δράσουμε και διαφορετικά οι πολυεθνικές στον τομέα της μεταποίησης τροφίμων και... Ε, θα πρέπει και αυτές να βοηθήσουν οι οποίες μέχρι τώρα έχουν ουσιαστικά καταστρέψει τις μικρές ε, επιχειρήσεις αλλά και τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις το ελεύθερο εμπόριο επίσης οι αρνητικές συνέπειες η ε, απερίμωση της υπαίθρου οφείλεται πολύ σε αυτά τα λυπηρά αποτελέσματα ε, στον τομέα της γεωργίας θα χρειαζόταν τεράστια χρήματα για να μπορέσουμε τεράστια ποσά για να μπορέσουμε ε, να, να αναστρέψουμε την κατάσταση. Λεπτό, παρακαλώ. Η κυρία Ντότς, για ένα λεπτό παρακαλώ. Η κυρία Ντότς, για ένα λεπτό. Uh, thank you. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κατά την Παγκόσμια Σύνοδο, ο Γενικός Γραμματέας Πάνκι Μουνή είπε ότι η επιστημική κρίση σήμερα είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει για αύριο, για το αύριο. 9 δις ε, θα είναι ο πληθυσμός ε, πολύ σύντομα κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει οι γεωργοί να παράγουν 70% παραπάνω τρόφιμα. Η Ιρλανδία δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί αλλά οι περισσότεροι πιστεύουν στην Ιρλανδία ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τους δημιουργεί πρόβλημα στην παραγωγή τροφίμων γιατί τους υποχρεώνει να εφαρμόζουν πάρα πολλούς κανονισμούς, να περνούν από φοβερή γραφειοκρατία, κάτι το οποίο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν, δεν υπάρχει επιζητιστικό ε, πρόβλημα. Επίσης επηρεάζονται και οι τιμές. Αν οι γεωργοί δεν υποστηρίζονται μέσω των άμεσων ενισχύσεων, τότε θα πρέπει να αυξηθεί πρέπει να η παραγωγή, αυξάνοντας παράλληλα βέβαια και το κόστος. Αυτό κατά τη γνώμη μου θα, θα ε, το, το πρόβλημα θα λυθεί μόνο εάν δίνουμε τη δυνατότητα στους γεωργούς να καλλιεργήσουν και αυτό θα έπρεπε να είναι μια βασική συνιστόσα της δουλειά μας, ειδικά όταν πρόκειται ε, να αναθεωρήσουμε την κοινή γεωργική πολιτική. Ευχαριστώ. το τώρα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι από τους συγγραφείς της ε, έκθεσης αυτής και ε, νομίζω ότι στο σημείο αυτό πρέπει να ευχαριστήσω όλους αυτούς που βοήθησαν ε, να φτιαχτεί το κείμενο αυτό για το οποίο δεν υπήρχαν τροπολογίες. Ε, είμαστε όλοι σύμφωνοι ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε την εξάλληψη της πείνας στον πλανήτη μας γιατί ήμουν υπεύθυνη και για σχετικά θέματα για την εμπιστοστική ασφάλεια και στην προηγούμενη θητεία και θα ήθελα να τονίσω κάτι το οποίο φαίνεται ότι το ξεχνάμε οι αγρότες είναι αυτοί που θρέφουν ουσιαστικά τον πλανήτη μας αν ο καιρός είναι καλός και μπορούν να παράγουν τα προϊόντα τους τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα θα πρέπει λοιπόν να χαράξουμε πολιτικές που θα επιτρέπουν στους αγρότες μας να παράγουν τρόφιμα θέλ, χρειάζονται αξιοπρεπείς τιμές και σταθερά εισοδήματα για να μπορέσουν να δουλέψουν οι άνθρωποι αυτοί. Η κρίση η οποία, την οποία διατρέχουμε δεν τους εξασφαλίζει τα πράγματα αυτά και δεν μπορούμε να δαιμονοποιούμε την κοινή αγροτική πολιτική. μερικά η μεταρρύθμιση της κοινή αγροτικής πολιτικής ήταν καλή και δίχως την ΚΑΠ θα είχαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ μεγαλύτερα προβλήματα από ό,τι έχουμε αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν δεχόμαστε λοιπόν τα καλά στοιχεία της ΚΑΠ και να ζητήσουμε και από τις αναπτυσσόμενες χώρες να ακολουθούν αντίστοιχους κανόνες. Δεν μπορούμε να ε, αφήνουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες να κάνουν ό,τι τους αρέσει. Κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνουμε σκληροί και με τους εαυτούς μας και με τις κυβερνήσεις μας και με τις άλλες χώρες. Ο Γκερέρο Σαλόμ για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρα. Κύριε Επίτροπε, ομό, ο κόσμος έχει να αντιμετωπίζει δύο πολύ σημαντικές προκλήσεις. Την ε, κλιματική αλλαγή και την πείνα και τη φτώχεια στον κόσμο. Ε, και ο Επίτροπος και άλλοι έδωσαν τα αριθμητικά στοιχεία που ε, προέκυψαν από την τελευταία σύνοδο κορυφής της ΦΑΟ. Ένα δις ανθρώπων υποφέρουν από πείνα, 40 εκατομμύρια πεθαίνουν από τις παρενέργειες της ε, φτώχειας. Η επιστηστική κρίση πρώτα και η οικονομική κρίση μετά μας απομακρύνει πολύ από τους στόχους της χιλιετίας. Όχι απλώς δεν τους πλησιάζουμε, αλλά απομακρυνόμαστε από αυτούς. Είναι μακροπρόθεσμη προσπάθεια. Παρ' όλα αυτά τις τελευταίες εβδομάδες λάβαμε ανησυχητικά νέα η αντίσταση των ε, μεγάλων ε, εκπομπέων ανθράκα να λάβουν αποφάσεις θαραλές στην Κοπενχάγη και ε, η άρνηση των όσων συμμετείχαν στη διάσκεψη της ΦΑΟ στη Ρώμη να αναλάβουν δεσμεύσεις μας δένουν τα χέρια. Έχουμε προοδεύσει ως ανθρώπινο είδος διότι είδαμε ποιες είναι οι προκλήσεις που είχαμε και πήραμε την τύχη στα χέρια μας. Αυτό συμβαίνει και τώρα. Ξέρουμε ε, ποια είναι η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε, αλλά δεν μπορούμε πια να αντιδράσουμε. Γι' αυτό υποστηρίζω την, το ψήφισμα αυτό που ζητεί από το Κοινοβούλιο δράση και άμεση δράση. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κέλλερ, για ένα λεπτό παρακαλώ. Thank you. Article... Ευχαριστώ. Το άρθρο τη 248 της Συνθήκης της λέει ότι ο βασικός στόχος Ευρωπαϊκής Ένωση ε, στην αναψυκτική πολιτική της ε, είναι η μείωση και εξάλληψη της φτώχεια και της πείνα. Η φτώχεια είναι βασικός λόγος για την πείνα. Το ίδιο άρθρο αναφέρει επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα λάβει υπόψη του στόχου αυτού σε άλλε πολιτικέ που μπορεί να επηρεάσουν τι αναπτυσσόμενες χώρες αλλά με τις ε, επιδοτήσεις στις εξαγωγές ε, ουσιαστικά καταστρέφει την κατάσταση στις ε, άλλες χώρες με την ενίσχυση της φτώχειας και της πείνας. Αν θέλουμε λοιπόν να είμαστε αποτελεσματικοί πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν δημιουργούμε εμπόδια από άλλες πολιτικές. Διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους της χιλιετίας και πρέπει να μην μας διαφεύγει αυτό όταν αναθεωρούμε και μεταρρυθμίζουμε με πολιτικές όπως η κοινή γεωργική πολιτική και η κοινή αλληλευτική πολιτική. Ευχαριστώ. Η κυρία Μακίνε θέλει να κάνει δικαίωμα της μπλε κάρτας. Έχετε το λόγο κύριε Μακίνε. like... Δεν είναι κίτρινη, μπλε είναι η κάρτα. Θα ήθελα να ρωτήσω για τις επιστροφές, τις εξαγωγές, τι ελέγχθη. Εγώ μίλησα για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ για το γαλακτοκομικό τομέα υπάρχουν ε, επιστροφές κατά την εξαγωγή και οι μόνοι που παραπονέθηκαν ήταν η Νέα Ζηλανδία. Δεν κατάλαβα πού είναι το πρόβλημα. Ε, η κυρία Κέλλερ θέλει να απαντήσει. Η κυρία Κέλλερ θέλει να απαντήσει. Yes, of course. Um, of course the frozen chicken example. Βέβαια, τα κατεψυγμένα κοτόπουλα που γνωρίζετε όλοι είναι ένα παράδειγμα, αλλά οι ντομάτε, για παράδειγμα, είναι επιδοτούμενε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με υψηλέ επιδοτήσει. Ε, Στι αφρικανικέ αγορέ όμω ε, τα τοπικά προϊόντα είναι, έχουν χαμηλότερε τιμέ και άλλα δημιουργούνται πολύ μεγάλα προβλήματα και νομίζω ότι πρέπει κάτι να κάνουμε γι' αυτό. Σα ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας. Έχει το λόγο τώρα ο κύριος Γκλατφέλντερ για δύο λεπτά παρακαλώ. A világban egyre több tudós állítja azt, hogy 2030-ra egy... Οι επιστήμονες λένε ότι στον κόσμο μας το 2030 θα υπάρχει η πετρελαϊκή κρίση, υδατική κρίση και διατροφική και επιστημιστική κρίση. Δεν ξέρω αν έχουν δίκιο ή όχι, αλλά εκείνο το οποίο είναι γεγονός είναι ότι αυξάνεται συνεχώς ο πληθυσμός του πλανήτη και σε μερικές δεκαετίες ε, ε, το 20% ε, περίπου, το 1 πέμπτο ε, αν θέλετε του πληθυσμού θα πεινάει η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει δράση πριν να συμβούν όλα αυτά. Ή έχουμε μια κοινή αγροτική πολιτική και η πείνα κυρίες και κύριοι δεν υπάρχει μόνο στην Αφρική. Υπάρχει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν ε, βεβαίως... Ε, ε, υπάρχουν βέβαια περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου η, ε, δεν υπάρχει πρόβλημα πείνας και και τα έξοδα για τα, τρόφιμα είναι γύρω στο 10% του εισοδήματος του πολίτη. Υπάρχουν όμως περιοχές στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία όπου το 50% των εσόδων των πολιτών πάνε για διατροφή. Θα πρέπει λοιπόν να καθίσουμε να τα σκεφτούμε αυτά και όταν φτιάχνουμε καινούριου κανονισμούς που ουσιαστικά αυξάνουν τις τιμές των τροφίμων ε, πρέπει να ε, προσέχουμε τι γίνεται και ποιες θα είναι οι συνέπειες. Δημιουργούμε, αν θέλετε, πείνα με ορισμένα πράγματα που κάνουμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση όταν θέλουμε να ε, να προστατεύσουμε τον πλανήτη, να μειώσουμε το ανθρακικό αποτύπωμα παραδείγματο χάρη τη παραγωγή κρέατο ή πουλερικών. σω κάνουμε ένα παιδί να πεινάει. subnutrite în trecut de ajungându-se la drama. Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα η κατάσταση είναι δραματική. Δυστυχώς, ε, Ακούσαμε ότι οι πλούσιες χώρες με πάρα πολύ κινησμό αντιμετώπισαν την ανάγκη της αντιμετώπισης του προβλήματος. Πολλά, πολλά, πολλοί αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων δεν πήγαν καν στην παγκόσμια διάσκεψη, εκτός από τον κύριο Μπερουσκόνη βέβαια. Και μιλάμε για χώρες ε, που είναι άνω του 60% του παγκόσμιου ΑΕΠ και που εκπροσωπούν το τραπεζικό σύστημα και βέβαια είναι πάρα πολύ μεγάλος ο κινησμός τους ε, απέναντι στις φτωχέ χώρες οι οποίες καθόλου υπεύθυνε δεν είναι για την ε, κατάσταση που αντιμετωπίζουν. Πολύ είναι η πείνα στον κόσμο. Από το 1970 Όλο και περισσότεροι είναι εκείνοι που πεθαίνουν από την πείνα. Μιλάμε για ανθρώπινη τραγωδία η οποία θα μας, επηρεάσει, θα μας ακόμη περισσότερο στο μέλλον και η κατάσταση θα γίνει πραγματικά τρομακτική. Εδώ και 20 χρόνια η επισητιστική κρίση σιγά σιγά άρχισε να συμβαίνει λόγω των πολιτικών μας. Το 2006 ε, στην Σύνοδο του ΦΑΟ διαπιστώσαμε φοβερή επιδείνωση της κατάστασης. Σήμερα μιλάμε για άνοιγμα των αγορών, ε, για την ε, διευκόλυνση, την ενίσχυση των γυναικών γεωργών, για την εξάλληψη της πίνης. Κρέτου, ο, ο συνάδελφος ο κύριος Στογιάνοφ θέλει να σας υποβάλει μια ερώτηση. Θέλετε να απαντήσετε. Θέλετε να απαντήσετε. Θέλετε να απαντήσετε σε ερώτηση που θα σας υποβάλει ο συνάδελφος, ο κ. Στογιάννοφ. Θέλετε να απαντήσετε στην ερώτηση που θα σας, υποβάλει ο συνάδελφος, ο κ. Στογιάννοφ. Λοιπόν, ε. Κύριε Στογιάννοφ, δεν θα μπορέσετε να κάνετε χρήση της ε, μπλε κάρτας. Συνεχίζουμε. Επόμενη ομιλήτρια, η κυρία Εράνς Γκαρσία, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να, συγχαρώ την κυρία Μαγκίνες για αυτή την πρωτοβουλία που καταδεικνύει το σημαντικό ρόλο της ε, κοινής αγροτικής πολιτικής εις ό,τι αφορά την επιστηστική ασφάλεια. Τώρα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να μειώσει το βάρος ε, της ε, ΚΑΠ στον ε, ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, θα πρέπει να πούμε ότι η ΚΑΠ δεν είναι προτεραιότητα, όμως η πιστική ασφαλεία είναι. Στις τελευταίες δεκαετίες είδαμε ότι ήταν εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να υπάρχει πλήρης επιστηστική ασφάλεια. η αγορά των διατροφικών προϊόντων δεν είναι σαν μια οποιοδήποτε άλλη. Ο, ο Γεωργός χρειάζεται την Ευρώπη και η Ευρώπη χρειάζεται τον Γεωργό. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε αλλαγή πορείας. Άμεσες ενισχύσεις στους Γεωργούς, πολιτική διαχείριση των γεωργικών αγορών, που να έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη σταθερότητα στι τιμές, κάτι που θα ήταν υποφελέ όχι μόνο για τους γεωργού, αλλά και για τους καταναλωτές και τις τρίτες χώρες. Απαραίτητο επίσης είναι να υπάρχουν βέλτιστες πρακτικές για να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των διαφόρων κρίκων της διατροφικής αλυσίδα να μην υπάρχουν καταχρήσει και να υπάρχει πιο δίκαια περιθώρια κέρδους στι στις επιχειρήσεις. Και βεβαίως μια ενημέρωση του πολίτη που θα πρέπει να γνωρίζει τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από βάση νομοθεσίας ε, σε όλα τα θέματα της ε, Γεωργίας. Διότι μην ξεχνάμε ότι οι Ευρωπαίοι Γεωργοί ανταγωνίζονται γεωργούς από τρίτες χώρες όπου τα πρότυπα είναι πολύ χαμηλότερα. Η παραγωγή αυτή των τρίτων χωρών προτιμούν να εξάγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρά να τροφοδοτούν τις αγορές των ειδικών τους χωρών. Για τον απλούστατο λόγο ότι είναι πολύ πιο αποδοτικό κάτι τέτοιο. Τελειώσαν εδώ οι παρεμβάσει των εγγεγραμμένων μελών και ερχόμαστε στη διαδικασία Catch the Eye. Το θέμα είναι πολύ ενδιαφέρον και έχουν ζητήσει το λόγο πολλοί συνάδελφοι. Κρατήστε σας παρακαλώ το χρόνο του ενός λεπτού γιατί είμαστε ήδη αργά. Ε, η κυρία Στρίφλερ έχει το λόγο πρώτη παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Είπαμε πριν από λίγο ότι κάθε, πέντε δευτερόλεπτα ένα παιδί πεθαίνει στον κόσμο από την πείνα και λέμε ότι πάνω από ένα δισεκατομμύριο είναι τα άτομα που δεν τρέφονται σωστά. Το ζήτημα της επιστημιστικής ασφάλειας είναι εξαιρετική σημασία, επίγουσα σημασία και πρέπει να είναι αντικείμενο πολιτικών και σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο. Ε, πρέπει να υπάρχει συντονισμός των πολιτικών ε, για την εστίαση στους στόχους της χιλιετίας. Ε, το 1 δισεκατομμύριο ευρώ είναι μια πρώτη, ένα πρώτο βήμα ώστε να επικεντρωθούμε στις ε, μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις, ε, στις οικογενειακές καλλιέργειες και ειδικότερα αυτές ε, τις οποίες καλλιεργούν γυναίκες και που πλήττονται περισσότερο από την κρίση. Η βιώσιμη γεωργία πρέπει να είναι προτεραιότητα, πρέπει να υπάρχει καινοτομία, όπως για παράδειγμα ένας φόρος που θα συνοδεύσει την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή ο κύριος Κόρτες Λάστρα για ένα λεπτό επίσης. <clears throat> Ευχαριστώ. Μετά την τελευταία διάσκεψη της ΦΑΟ θα ήθελα να εκφράσω την απογοήτευσή μου για την κοινωνική, ε, επικοινωνιακή ε, και στρατηγική αποτυχία γιατί δεν ε, εξευρεθεί συμφωνία για την ενίσχυση των ε, φτωχών. Όλα μείναν όπως είχαν. Όταν μιλάμε για αυτά τα θέματα, πολύ συχνά ξεχνάμε το θέμα του νερού, της σπάνιδος του ύδατος. Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής και οικονομικής κλίσης που μας πληττεί, θέλουμε δέσμευση από τις αναπτυσσόμενες χώρες για τη δημιουργία ενός διεθνούς φόρουμ περισυλλογής για το θέμα του ύδατος που είναι το πολυτιμότερο δημόσιο αγαθό. Αν δεν φροντίσουμε το νερό θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Στην Αγγλία του 18ου αιώνα ο Τόμας Μάουθα είχε ήδη προβλέψει ορισμένα προβλήματα σχετικά με την διατροφική ε, επάρκεια. Βέβαια έκτοτε έγιναν, έγινε βιομηχανική επανάσταση κτλ. Αλλά ε, ε, ε, σε πολλά πράγματα βγήκε και αληθινός γιατί έχει τριπλασιαστεί ο πληθυσμός και είναι πολύ μεγάλος ο ρυθμός των ανθρώπων που πεινούν πρέπει λοιπόν για να μπορέσουμε να ε, εξαλείψουμε την πείνα για τους ανθρώπους αυτούς και να βοηθήσουμε να σώσουμε ουσιαστικά τις ζωές των παιδιών και των νέων να αυξήσουμε την παραγωγικότητα στον αγροτικό τομέα. Εκείνο το οποίο κάνουμε εδώ όμως στην Ευρώπη ε, ε, τα, τα προβλήματα δεν τα αντιμετωπίσαμε και συνεχίζουμε να τρώμε κρέας. Mr. Jakob, please. Ich habe meinen Namen akustisch nicht verstanden. Συγγνώμη, δεν είχα ακούσει το όνομά μου. το δικαίωμα για την διατροφή είναι ανθρώπινο δικαίωμα και τα επιστημονικά στοιχεία που έχουμε ε, μας λένε ότι η αύξηση του πληθυσμού θα οδηγήσει όλο και περισσότερο αριθμό ανθρώπων στην πείνα. Για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε λοιπόν το πρόβλημα πρέπει να κάνουμε ορισμένα πράγματα. Πρώτα πρώτα στις αναπτυσσόμενες χώρες να υπάρχουν δημοκρατικές δομές. Δεύτερον, κατά καταπολέμηση της διαφοράς. Τρίτον, στις αναπτυσσόμενες χώρες ε, καλύτερη γεωργία και ε, αγορές και μετά έρχονται οι επενδύσεις. Τα τρία πρώτα θέματα δεν τα συζητούμε και πολύ και επιμένουμε στο θέμα των επενδύσεων και έτσι πηγαίνουν χρήματα σε λάθος περιοχές. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συνεχίσω αυτό που είχα πει προχθές και μίλησε ειδικότερα για την Αφρική και την έλλειψη υποστήριξης από τις πιο βιομηχανοποιημένες χώρες σε σχέση με την επιστημιστική κρίση. Επειδή λοιπόν έγινε η παγκόσμια διάσκεψη στο, του ΦΑΟ, οι πολλοί, πολλοί κατηγόρησαν τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις για αρπαγή γεών πάνω από 40 από τις, από τις ότι υπήρχε τάση από πολλές πλούσιες χώρες να χρησιμοποιούν χημικά λιπάσματα ε, αντί να ε, ενθαρρύνουν τις βιώσιμες, τις βιώσιμες καλλιέργειες ε, και ε, την έλλειψη αγροπεριβαλλοντικών μέτρων. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια παγκόσμια εταιρική σχέση για την καταπολέμηση της ένδυας και της φτώχειας προς αυτή την κατεύθυνση. Μου λένε ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η κυρία Κόστιγκερ έχει το λόγο τώρα για ένα λεπτό. Mrs. Köstinger. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε μακροπρόθεσμη επιστημιστική ασφάλεια είναι ο βασικός στόχος της κοινή αγροτικής πολιτικής. Είναι, ε, ε, αν θέλουμε στο μέλλον να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε τις προκλήσεις που θα ε, βρούμε μπροστά μας πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό και ένα βασικό στοιχείο της επιστημιστικής ασφάλειας στην Ευρώπη είναι ε, και η ε, σχέση μας, η διατήρηση κάποιων οικοσυστημάτων και η σχέση σωστή με τις ε, τρίτες χώρες. Η διεθνή συνεργασία για την επιστημιστική ασφάλεια είναι απαραίτητη. Είναι και δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να δράμε μονομένα. Ζούμε σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Λόγο τώρα για ένα λεπτό Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς, ενδεχομένως να επαναλάβω κάτι το οποίο είπε συνάδελφος προηγουμένως. Θα ήθελα να πω ότι με καταθλίβει το γεγονός ότι έχουμε τόσες καλλιέργητες εκτάσεις ε, στην Ευρώπη και καταγγέλουμε παράλληλα ε, την πείνα ε, στον κόσμο. Και ο Επίτροπος μίλησε για αυτό το θέμα. Δηλαδή ο κίνδυνος για τον κίνδυνο που μπορεί να υπάρχει μέσω της ε, έλλειψης αυτάρκειας. Δεν είναι το ίδιο πράγμα αυτό με την επιστημιστική ασφάλεια. Ε, η κλιματική αλλαγή έχει διαφορετικό αποτέλεσμα σε κάθε ε, περιοχή. Κάτι που σημαίνει ότι ένας, μια χώρα μπορεί να μπορεί να παράγει αυτό που χρειάζεται. Κυρία Χάρκιν, ευχαριστώ πρόεδρε. Πρώτα-πρώτα η σχέση μεταξύ κλιματική αλλαγή και πείνας, όπως είπε και ο Μπανκιμούν στην ε, Ρώμη μέχρι το 2050 τότε θα πρέπει λόγω των καινούριων κλιματικών συνθήκων να παράγουμε 70% παραπάνω ε, τρόφιμα είναι όντως υπάρχει μεγάλη σχέση μεταξύ πείνας, τόχες αύξηση του πληθυσμού και κλιματικής αλλαγής. Από εκεί και πέρα βεβαίως η εύκολη λύση είναι να επιτιθέμεθα στην ΚΑΠ αλλά η ΚΑΠ μεταρρυθμίστηκε και δεν νομίζω ότι ε, αλλά δεν νομίζω ότι είναι σωστό αυτό. Παραδείγματος χάρη για την βιομηχανία ζάχαρης στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία ουσιαστικά διαλύθηκε, καταστράφηκε με την τελευταία μεταρρύθμιση ε, βόηθησε αυτό τις αναπτυσσόμενες χώρες δεν θέλω να ελαχιστοποιήσω και να αγνοήσω το πρόβλημα της παγκόσμιας πείνας αλλά θα πρέπει να τα δούμε τα πράγματα πιο λογικά Ευχαριστώ. ευχαριστώ, On erittäin Kööpenhaminan ilmastokokouksen Ευχαριστώ. Ε, είναι καλό το ότι συσχετίζουμε με την κλιματική αλλαγή το θέμα αυτό, όταν το ότι συζητούμε δηλαδή παράλληλα το θέμα της επιστημικής ασφάλειας και της κλιματικής μεταβολής, γιατί υπάρχει όντως μία σχέση. Έχουμε κάποιους στόχους για τα βιοκαύσιμα, για παράδειγμα, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα έχουμε χρησιμοποιήσει πάρα πολλές εκτάσεις για την ύπαρξη εγκαταστάσεων βιοκαυσίμων. Και στην κοινή γεωργική πολιτική υπήρξαν πολλές τρευλώσεις. Κάναμε εξαγωγή του πλεονάσματός μας στις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι και σήμερα ακόμα έχουμε πολλά τρόφιμα στον κόσμο, έχουμε επαρκή τρόφιμα, αλλά δεν έχουμε το, την θέληση να τα κατανείμουμε. Κέρσκι παρακαλώ pani przewodnicząca! szanowni państwo! na ostatnim szczycie fao państwa nie Κατά τη διάρκεια της τελευταίας ε, παγκόσμιας ε, συνόδου, τα κράτη-μέλη δεν μπορούσαν να καταλήξουν σε μία λογική πρόταση. Η έλλειψη διεθνούς στρατηγικής είναι κάτι το ανησυχητικό. Αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι θα αυξηθεί σε πάνω από 9 δις πληθυσμός μέχρι το 2020, 15. Ε, Όταν ε, βλέπουμε και την αύξηση των τιμών των τροφίμων, μπορούμε να φανταστούμε την ε, απειλή της, του θανάτου από την πείνα για πάρα πολλούς ανθρώπους. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε όλες αυτές τις, όλες αυτές τις δράσεις που μπορούν να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά και να δούμε βέβαια και τις τάσεις που υπάρχουν στις διεθνείς αγορές. Περιορισμό τη κοινή γεωργική πολιτική νομίζω ότι δεν έχει νόημα γιατί δημιουργεί πρόβλημα και απειλή στην επιστημιστική μας ε, ασφάλεια. Πρέπει να βοηθήσουμε τι αναπτυσσόμενες χώρες να έχουν τέτοια γεωργική πολιτική που μπορούν, που να του επιτρέπει αυτάρκεια. Ευχαριστώ. Η συζήτηση θα κλείσει ο κύριο Επίτροπο. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Και εγώ λυπούμε βαθιά που κανένας από τους ηγέτες της ομάδας των 8 δεν ήταν παρόν. Ο πρώτος Μπαρόζο Ήτο. Και η απουσία των ηγετών επέτεινε την εντύπωση που είχαμε για αποτυχία. Είναι πολύ σημαντικό όμως να έχουμε υπόψη ότι καταφέραμε να διατηρήσουμε το θέμα στην πολιτική ατζέντα. Και οι δύο διασκέψεις του 2009 το απέδειξαν αυτό. Όποτε συναντώνται οι ηγέτες, η ομάδα των 20 στο Πίτσμπεργκ μίλησε για την ε, αναπτυξιακή συνεργασία και την αναπτυξιακή πολιτική. Αυτή είναι μια θετική εξέλιξη. Ήμουν στη Ρώμη και εκτός από την οριστική δήλωση που συμφωνώ ήταν κάπως απογοητευτική, οι συζητήσεις ήταν χρήσιμες, καλές και νομίζω ότι κάτι μπορεί να προκύψει. Η συζήτηση ας πούμε για την πώληση γόνιμων γεών στις αναπτυσσόμενες χώρες. Χώρες που δεν έχουν δηλαδή γόνιμες γες να αγοράσουν τέτοιες από άλλες αναπτυσσόμενες χώρες. Νέες ιδέες λοιπόν έχουν τεθεί επιτάπητος. Τώρα, για την ΚΑΠ δεν είναι ιδεώδης. Τίποτα εξάλλου δεν είναι στον κόσμο τούτο τα αποτελέσματα της κοινή αγροτικής πολιτικής στον αναπτυσσόμενο κόσμο πιστεύω ότι ήταν τα λιγότερο επιζήμια. Δηλαδή από τις πρακτικές των άλλων μεγάλων δυνάμεων η ευρωπαϊκή κοινή αγροτική πολιτική ήταν η ο λιγότερο επιζήμια για να το θέσουμε ένα σχήμα λιτότητος εμπορικές πολιτικές άλλων οικονομικών σχηματισμών έχουν ζημιώσει περισσότερο τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Είμαι και κάπως απογοητευμένος γιατί ποτέ δεν είμαστε ικανοποιημένοι στην Ευρώπη με την επιστηστική βοήθεια κάναμε ένα πολύ μεγάλο βήμα προς τα μπρος. Ένα δις ευρώ. Δεν παρέχει τρόφιμο, έτοιμη τροφή, αλλά σπόρους προς καλλιέργεια και βοήθεια προς τους μικρούς γεωργούς του αναπτυσσομένου κόσμου. Αυτό είναι μεγάλη καινοτομία, πολύ θετική, που έχει αναγνωριστεί ως τέτοια και από την Παγκόσμια Τράπεζα, που έχει ασπαστεί τον μηχανισμό. Δεν θα πρέπει λοιπόν πάντα να αυτομαστιγωνόμαστε στην Ευρώπη. Σε αυτό που διαφωνώ με τον προκατοχό μου, με αυτό που διαφωνώ και με αυτό που είπε ο κύριος που έχει αποχωρήσει τώρα, ο κύριος Λε Ιαρίκ. Κάποιος είπε ότι είναι σοσιαλιστής. Όχι, κομμουνιστής είναι ο άνθρωπος. Γι' αυτό λέει τα πράγματα που λέει. Στη Λάκουιλα τώρα. <coughs> Υποσχεθήκαμε δις δολαριών. Και έτσι είμαστε μακράν ο μεγαλύτερος δωρητής στην παγκόσμια σκηνή. Και θα τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας αυτές. Και αυτό το 20% που έχουμε πει ότι θα απελευθερώσουμε από αυτό το κοντήλιο θα το κάνουμε στον τον πιο σύντομα. Ένα τελευταίο, αν μου επιτρέπετε πρόεδρε, για το πρόγραμμα εργασία του 2010. Η Κομισιόν θα παρουσιάσει στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο μια ανακοίνωση για τη νέα, την ανανεωμένη πολιτική για την επιστηστική ασφάλεια, τη διατροφή, την ποιότητα των τροφίμων, την κοινωνική προστασία και κοινωνική πολιτική, τις συνέπειες των βιοκαυσίμων στην παραγωγή στην γεωργία, τις νέες τεχνολογίες και πολλά άλλα. Η ανακοίνωση ο στόχο θα έχει ένα Ανανέωση της δεσμευσής μας να βοηθήσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες στην γεωργική τους παραγωγή. Ιδιαίτερα λόγω της συνεχόμενης αύξησης ε, του πληθυσμού και των ε, στόχων που έχουμε για βιώσιμη γεωργική παραγωγή. 2. Να ξεκινήσει μια περισυλλογή για το πώς η Ένωση μπορεί να υποστηρίξει νομοθετικά και στρατηγικά αυτές τις νέες πολιτικές. Τρία. να εφαρμόσουμε τα συμπεράσματα της άκρα. Τέσσερα. Πώς θα επιταχύνουμε τη διαδικασία των MDG και ιδιαίτερα του MDG1. Πέντε. Να καθορίσουμε τη θέση μας έναντι των τελευταίων εξελίξεων και έξι επιστηστική ασφάλεια. Θα γίνει ευρία διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερομένους και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι με την ανακοίνωσή μας αυτή. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω λάβει έξι προτάσεις ψηφίσματος σχετικά με το θέμα της συζήτησης, επί των οποίων η ψηφοφορία θα γίνει αύριο. Το θέμα έληξε λοιπόν, η συζήτηση αυτή έληξε. Και ερχόμαστε ε, στο επόμενο θέμα της ημερήσιάς μας διάταξης που προβλέπει τη δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τις εισαγωγές κρέατος προέλευσης τρίτων χωρών. Θα ξεκινήσουμε με την Επίτροπο την κυρία Βασιλείου. Έχετε το λόγο κυρία Επίτροπο. Ε,